Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τους ε, εισηγητές ε, για τη συνεργασία τους. Είμαστε ευτυχείς που βρήκαμε πραγματικά ένα πεδίο συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό δια, Σταθερότητας. Νομίζω ότι οι συμβιβαστικές προτάσεις σε συνεργασία με τους σκιώδεις καλύπτουν τους πιο σημαντικούς τομείς γύρω από τα θέματα της ε, διαφοροποιούμενης ή μεταβλητής ολοκλήρωσης, της διεύρυνσης και της γενικότερης ολοκλήρωσης στο εσωτερικό της Ένωσης σε σχέση με τις προσπάθειες των κρατών μελών για την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική σύγκληση. Από τη μία υπογραμμίζουμε ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η καλύτερη για την λειτουργία της Ένωσης και έτσι η προσαρμογή και η ανανέωση ε, της πολιτικής αυτής ε, φέρνει στην επικαιρότητα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων με στόχο την ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα των κοινοτικών πολιτικών. Τώρα σχετικά για την, με την Τραπεζική Ένωση, οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση θα πρέπει να συνεχιστούν. Πρέπει να ενθαρρύνουμε φυσικά α, και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί από ορισμένα κράτη-μέλη έτσι ώστε να προωθήσουν τη σύνδεσή τους. Και εδώ τίθεται το θέμα και του σωστού συνδυασμού των διαφθρωτικών ταμείων, του αναπτυξιακών μέσων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να υπάρξει σωστός συντονισμός και τέλος να προσθέσω ότι δυστυχώς η λεγόμενη αυτή διαφοροποιούμενη ολοκλήρωση ή μεταβλητή ολοκλήρωση στην ουσία γίνεται αντιληπτή σαν κάτι το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας μελών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμποδίζοντας να υπάρξει μια σωστή πολιτική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, η οποία είναι απαραίτητη για να καταλήξουμε σε μια όλο ένα πιο στενή ένωση. Η μη συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας στο χώρο Σέγγεν Φοβάμαι ότι θα εμβαθύνει αυτή την αίσθηση διάκρισης ιδιαίτερα στις χώρες που πρόσφατα έγιναν μέλη. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά συνάδελφοι και περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμασούρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο έχει ενημερώσει το σύνολο των πολιτικών ομάδων και έχει καταλήξει σε συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες είναι αποδεκτές από όλους. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμφωνούμε με τη βασική ανησυχία την οποία έχει εκφράσει ο κ. Φοντζούλητσα ότι δηλαδή αν εμείς θέλουμε να προωθήσουμε τις λεγόμενες διαφοροποιούμενες μορφές ολοκλήρωσης και συνεργασίας, σε πολιτικό επίπεδο δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε δύο κατηγορίες μελών. Δεν αναφέρομαι σε καλούς κακούς μαθητές. Υπάρχουν κάποιοι τομείς για τους οποίους υπάρχουν φυσικά διαφορετικές συνθήκες Υπάρχει και διαφορετική βούληση, αυτό ποικίλει ανάλογα με το θέμα, ας πούμε ενισχυμένη συνεργασία, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα οι ίδιες χώρες αυτές οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν ακόμα περισσότερο και να έχουν μια πιο ενισχυμένη μορφή συνεργασίας στον ένα τομέα και λιγότερο στον άλλο. Ο εισηγητής έχει λάβει υπόψη πολλές από τις τροπολογίες μας και τον ευχαριστούμε. Υπάρχει ένα θέμα πάνω στο οποίο δεν καταλήξαμε σε συμβιβαστική. Είναι το «ή» αγγλικό. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επιθυμεί πάντα να υπάρξει αναφορά στο μέσο α, α, τεχνικής ενίσχυσης τεχνικής στήριξης. Ε, είναι κάτι το οποίο ανήκει, θα έλεγα, στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω να συμφωνήσουμε σε αυτό, γιατί αλλιώς θα τηρήσουμε στάση αποχής σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ. Σταμπάτη για τους συντηρητικούς. Κυρία Πρόεδρε, είναι μέθοδος ολοκλήρωσης να προχωρούν κάποιες χώρες, να βολιδοσκοπούν το έδαφος και να συμπαρασύρουν άλλες. Είναι η ολοκλήρωση δύο ταχυτήτων. Μπορεί να έχει νόημα κάτι τέτοιο. Εκτός και άλλοι, αν κάποιοι τολμήσουν να αποσυνδεθούν από την ολοκλήρωση. Αυτό δεν είναι επιθυμητό. Η ιδέα είναι να δοκιμάσουν καταρχήν κάποιες χώρες που θα είναι φυλακή. εάν προχωρεί το σύστημα και είναι λειτουργικό. Και αυτό είναι ένα σύστημα που στηρίζει η ομάδα μας. Αλλά έχουμε την εντύπωση ότι εδώ δεν πρόκειται για μεταβλητή ολοκλήρωση, αλλά ε, για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις της ε, συγκέντρωσης συγκεντρωποίησης. Δηλαδή διαφαίνονται τέτοιες τάσεις περαιτέρω συγκέντρωσης και η ομάδα των συντηρητικών δεν μπορεί να συμφωνήσει με κάτι τέτοιο. Εδώ αναφέρεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο EMSM, ο οποίος ε, δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίζει προβλήματα, κρίσεις ε, ή να παρεμβαίνει όταν διατρέχει κίνδυνο το ευρώ. Αυτή ήταν η ιδέα. Και τα κράτη-μέλη ε, συνεισέφεραν σε αυτόν τον μηχανισμό και βέβαια τα κράτη-μέλη φροντίζουν, και είναι λογικό αυτό, να ε, χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που έχουν διαθέσει για την Ευρώπη. Οπότε εδώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για περαιτέρω συγκέντρωση, δεν είναι αυτό το νόημα της όλης, του όλου εγχειρήματο και ο υπουργό Οικονομικών μας ε, είχε πει και στο Κοινοβούλιο σαφώς ε, ότι μια αλλαγή του ESM προς ε, την περαιτέρω συγκέντρωση και ενίσχυση Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων δεν τον βρίσκει σύμφωνο. Και εμείς πιστεύουμε ότι δεν πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση όπου θα ε, φέρομαι και άλλα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στο εγχείρημα της περαιτέρω συγκέντρωσης, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να περιμένουν ε, και να δουν, να έχουν δηλαδή ένα περιθώριο ε, αναμονής. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Σταρμπάτη, η κυρία Βίρινγκ για την ομάδα των φιλελευθέρων. Ε, αγαπητέ κύριε Φρουντζουλίκ, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για την ε, συνεργασία και το καλό αποτέλεσμα. Με χαρά επιβεβαιώνω ότι ε, λήφθησαν υπόψη οι απόψεις μας στις συμβιβαστικές. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να τις στηρίξουμε όλες. Οι αλλαγές τελευταία στιγμής στη συμβιβαστική ή e, δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, δεν θα την ψηφίσουμε. Τονίζω για το μέλλον το εξής. Μην κάνετε αλλαγές τελευταία στιγμή σε κάτι που έχει συμφωνηθεί ήδη από όλους. Οι συμβιβαστικέ που στηρίζομαι δείχνουν ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η σωστή. Απαιτεί περισσότερη ολοκληρωμένη νομισματική ένωση, πιο ανθεκτική τραπεζική ένωση και βελτιώνει την δημοκρατική λογοδοσία στην οικονομική διακυβέρνηση. Το κείμενο ζητάει μια ισχυρότερη ένωση, μια περισσότερο ολοκληρωμένη ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίρινγκ. Για τους πρασίνους, δεν, από τους πρασίνους δεν έχουμε σήμερα κανέναν. Για την ομάδα Γκουε ο κύριος Σίρντεβαν δεν είναι εδώ. Άλλος κανείς θα μιλήσει για την Γκουε. Όχι. Για την EFDD Κανείς επίσης. Η ομάδα ΙΕΝΕΦ, e όχι, δεν υπάρχει κανείς, οπότε πάμε στο Catch the Eye και η κυρία Περέ ζήτησε το λόγο. Είναι λίγο αργά, επειδή θα ψηφίσουμε έτσι καλλιώς σε λίγο και ξέρουν όλοι πολύ καλά τι τροπολογίες έχω υποβάλει. Όμως το κείμενο προδικάζει στη συμβαστική C ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αναφέρει το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Το Ευρωπαϊκό... Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να πούμε στη συμβαστική ως προς την δημιουργία ενός διαδόχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, διότι κανείς δεν γνωρίζει ε, ποιο θα είναι αυτό το πρόγραμμα ή που θα διαδεχθεί. Um λοιπόν, κοιτάζω να δω αν ζητεί άλλο το λόγο στα πλαίσια του Catch the Eye. Δεν βλέπω κανέναν, άρα δίνω το λόγο στον κύριο εισηγητή, τον κύριο Φρουντσουλίκα. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις ε, παρεμβάσεις τους. Ωστόσο, από το συνάδελφο Λαμασούρ, καταλαβαίνω ότι απλώς θα απόσχουν από την ε, συμβαστική που ανέφερε και ο κ. Λαμασούρ, αλλά θα υπερψηφιστεί η έκθεση από την ομάδα του. Για άλλη μια φορά, για όλους, είναι σημαντικό να οδηγηθούμε προς ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικό είναι αυτή η Τραπεζική Ένωση να γίνει επιτέλου πραγματικότητα. Όλοι το επιθυμούν και είναι αρκετά σημαντικό και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν. Και στην Ευρωζώνη βεβαίως. Ωστόσο, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι μου απέστειλαν email λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος Υπάρχει απειλή ε, εάν δημιουργήσουμε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για την ε, συνεργασία σας. Ε, hierfür später werden wir dann auch noch... Αργότερα θα ψηφίσουμε. Σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης κοινέ διατάξει για 7 ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, το Κοινωνικό, το Ταμείο Συνοχής, της θάλασσα και της Αλληλεία, για το άσυλο και τη μετανάστευση εσωτερική ασφάλεια και διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων. Μεγάλο βήμα για ένα σημαντικό θέμα. Η κυρία Μάλετιτς δεν είναι εδώ η από το ΕΛΚ. Ο κύριος Φέρμπερ, ο Μάρκος Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με, για τις κοινέ διατάξεις συνενώνει 7 ευρωπαϊκά ταμεία. Ε, ο στόχος είναι κοινοί απλωστευμένοι κανόνες που θα μειώνουν τη διοικητική επιβάρυνση για τις αρχές και τους δικαιούχους. 142 ε, τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Πολλές δεν μπορούν να περάσουν σε συμβιβαστικέ. Πρέπει να ψηφίσουμε μία προς μία εκεί. 15 ε, τροπολογίες υπάρχουν μόνο για το 160 για το τερματισμό των συντελεστών συγχρηματοδότησης. Αυτό έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Ρέτζιο Επαρκώς. Δεν ξέρω αν η γνωμοδότησή μας θα ληφθεί υπόψη εδώ. Στη συνάντηση των σχεδόν συμφωνήσαμε ότι επειδή ε, οι τροπολογίες πρότειναν ε, αλλαγές εκτός πεδίου ε, Οικονομικής Επιτροπής σκεφτήκαμε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή σε βασικά θέματα για τα οποία είμαστε αρμόδιοι. Ε, το άρθρο 10 για τα ταμεία ε, διαρθρωτικά και επενδυτικά, για την ε, μακροερασιμότητα, εκεί έχουμε, είχαμε αρχικά 142 και τις μειώσαμε. Θέλουμε να συμφωνήσουμε για το άρθρο 15. Η πρόταση της Κομισιόν για τη μακροοικονομική ερασιμότητα Μοιάζει ενοιολογικά με την δημοσιονομική περίοδο την κοινή. Βλέπουμε ότι το ΕΛΚ, οι Φιλελεύθεροι και οι ΕΣΥΑΡ στηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν με κάποιες αλλαγές και οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν νέα λύση η οποία είχε προετοιμαστεί και στην Επιτροπή Ρέτζη. Κάποιοι από Γκουε και SND θέλουν να καταργηθεί το 2015. Εμείς δεν προσπαθούμε να βρούμε λύση συμβιβαστική έχοντας υπόψη την ανάγκη να συνδέσουμε τις μεταρρυθμίσεις με τις επενδύσεις και την χρηστή διακυβέρνηση για να έχουμε αποτελέσματα. Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών, ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργία απασχόλησης, ε, ε θέσεων εργασίας. Θέλουμε να ευχαριστούμε όλους τις, ε, ε, όσους συνεργάστηκαν και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συμβιβαστική λύση. Ε, στις 21 Νοεμβρίου ε, θα γίνει η ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο σκιώδης των Σοσιαλιστών δεν είναι εδώ. Ο κύριος Φεραραντίνο, παρακαλώ. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Χαίρετε, ο κύριος Κοτσολίνο δεν μπορεί να είναι εδώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αλλά μου ζήτησε να διαβάσω την εξής παρέμβαση. Θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου μου, ιδίω την εισηγήτρια Μάλετιτ, οι οποίοι όλοι μαζί συνεισέφεραν στο να εξετάσει σωστά η Επιτροπή ΕΚΟΝ το όλο θέμα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να σταθώ σε τρεις πτυχές. Πρώτον, θέλω να επικεντρωθώ στο πλέον αμφιλεγόμενο θέμα, το άρθρο 15 την οικονομική διακυβέρνηση. Εκεί όπου οι τροπολογίε των ομάδων συγκλίνουν, ιδίω ό,τι αφορά την μακροοικονομική ρεσιμότητα. Εδώ Θέλω να υπογραμμίσω ότι η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών υπέβαλε πολλαπλέ τροπολογίε που οδεύουν στην ίδια κατεύθυνση. Διαγράφεται η ουσία τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα κυρίω. Πρόκειται για μια πολιτική θέση που συνάδει με όσα είχαμε υποστηρίξει στι προηγούμενε ε, διαπραγματεύσει σε σχέση και με το κοινό, με το το που δω που. Θα πρέπει λοιπόν το, το όργανο αυτό να μην είναι περιτά τιμωρητικό και να μην τιμωρούνται οι διάφορες περιοχές για ευθύνες που δεν είναι δικές τους. Δεν θα πρέπει να πλήττονται όσοι κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν ο αδύναμος κρίκος, οι επενδύσεις. Ιδίω στρατηγικές επενδύσεις που ε, επιτρέπουν στο σύστημα να είναι ανθεκτικό και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας για μεγάλο διάστημα. Ήταν η μοναδική η ευκαιρία να ε, υλοποιηθεί το εργαλείο αυτό ε, το 2016 κατά της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Και τότε η προσπάθεια αυτή της Επιτροπής ε, κατέρευσε, επειδή ήταν προφανές ότι ήταν περιτά τα τιμωρητικά μέτρα. Επιπλέον, σε εκείνη την περίπτωση έγινε σαφές ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα δεν μπορεί να είναι μια δαμοκλειοσπάθη που θα λειτουργεί ω απειλή πάνω από τα κεφάλια των κρατών μελών ε, για να επηρεάζει και τι επιλογέ του και τι εσωτερικέ του ε, πολιτικέ. Πραγματικά αναρωτιέμαι και ρωτώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ γίνεται να σκεφτείτε ότι μπορεί να διακοπεί η πολιτική συνοχή σε μια διαδικασία για το έλλειμμα ε, υπέρμετρη και υπερβολική και χωρί να λάβετε υπόψη όλα τα άλλα μέτρα εφαρμογή τη μακρονομική αιρεσιμότητα, μεταξύ των οποίων οι διαδικασίε που μπορεί να επιβληθούν όπω πρόστιμα. Πραγματικά λυπούμε που πρέπει να διαπιστώσω ότι για το ίδιο θέμα υποβλήθηκαν και τροπολογίε που πηγαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Ε, υπ' αυτήν την έννοια ε, υπάρχουν και τροπολογίε που είναι τελείω αντίθετε με τι δικέ μα θέσει και θα έλεγα και με την ε, κοινή λογική που θα έπρεπε να μα έχει κάνει να έχουμε η κοινή μα εμπειρία. Τροπολογίε που ζητούν διαδεργαφή δυνατότητα ε, αναστολή τέτοιε διακασίε σε περίπτωση, που, σε περίπτωση έκτακτων οικονομικών συνθήκων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φεραντίνο. Ο κύριος Όσοκ, κανονικά θα έπρεπε να είναι το ECR, ο κύριος Σταρμπάτη. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Όσοκ ζητεί συγγνώμη και με παρακάλεσε να παρουσιάσω το κείμενό του εγώ. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να κάνουμε σχόλια για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για τη γνωμοδότηση. Όπως γνωρίζετε, το ECR χαιρετίζει τους κανόνες για τη ρύθμιση 7 Ευρωπαϊκών Ταμείων ε, υπό επιμερισμένη διαχείριση για ε, και ενοποιημένους κανόνες με μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις αρχές του προγρά... των προγραμμάτων και τους δικαιούχους. Προκειμένου περί των συγκεκριμένων τροπολογιών, το βασικό θέμα που μας χωρίζει στο άρθρο 15, είναι το άρθρο 15 και πώς να αντιμετωπίσουμε τις αναστολές πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων στα πλαίσια της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης. Προσπαθήσαμε να καταθέσουμε τροποποιητικές προτάσεις για, κατα, απαλήφοντας όλο το άρθρο αφενός και αφετέρου κάνοντας ε, την ε, ρυθμίζοντας το θέμα της αναστολής. Πιστεύω ότι θα πρέπει σε αυτό το θέμα να κρατήσουμε το κείμενο της Κομισιόν γιατί θεσπίζει διατάξεις που ήδη είχαν εισαχθεί και καταξιωθεί στην πράξη στα πλαίσια του τωρινού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. επιπλέον, το ECR δεν μπορεί να στηρίξει τροπολογίες που περιορίζουν το ρόλο του Συμβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, στηρίζομαι όμως τις προτάσεις του εισηγητή να ε, εισαγάγει μια ρήτρα διεξόδου ώστε η Κομισιόν να ε, κάνει σύσταση στο Συμβούλιο σχετικά με την ακύρωση της αναστολής σε περίπτωση εξαιρετικών οικονομικών περιστάσεων ή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του οικείου κράτους μέλους. Προκειμένου περί των άλλων θεμάτων, το ECR είναι κατά των τροπολογιών που ζητούν ιεράρχηση δηλαδή τον καθορισμό προτεραιοτήτων δυσκολεύομαι να πω τη λέξη mm. prioritization ε, πρόκειται για τα προγράμματα που αφορούν τη μετανάστευση, τα θέματα μετανάστευσης. Η σωστή χρηματοδότηση για αυτούς τους στόχους πρέπει να προβλέπεται μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Από την άλλη πλευρά στηρίζομαι τις τροπολογίες που ενδυναμώνουν την συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, κυρίως ε, μέσω των κυβερνήσεων. Επίσης, ε, συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι η πιο ε, στενή σύνδεση του CPR με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμεινού δηλαδή, θα έχει φέρει προστιθέμενη αξία και είμαστε κατά των τροπολογιών που υπονομεύουν αυτή τη σύνδεση. Γιατί, ε, ε, ευχαριστώ κύριε Σαρμπάτη, ο κύριος Τρεμόζα για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πλευράς φιλελευθέρων θεωρούμε ότι ο κανονισμός αυτός για τις κοινέ διατάξεις έχει σαν στόχο τη μείωση των αδικαιολόγητων γραφειοκρατικών εμποδίων. Θεωρούμε ότι η ευελιξία και η αποδοτικότητα είναι βασικός στόχος της πρότασης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μάλλον από τα κράτη-μέλη τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών διοικήσεων τους. Δεν έχει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρωτικές γραφειοκρατικές δομές και γι' αυτό έχουμε καταθέσει τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Η φιλελεύθεροι μέχρι τώρα ήταν υπέρ της αιρεσιμότητας που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές. Οι φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι οι αναχώρες τα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Είδαμε τις συμβιβαστικές προτάσεις των εισηγητών και ιδιαίτερα το ή αγγλικό δεν κατανοούμε γιατί κάποιες ομάδες αποφάσισαν να μην συμφωνήσουν στις συμβιβαστικές προτάσεις, εκεί που είναι τουλάχιστον δυνατό. Σχετικά με το άρθρο 15 που είναι αμφιλεγόμενο, σχετικά με την διακοπή της χρηματοδότησης αν υπάρχει σημαντική παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Νομίζω ότι το μέτρο αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει τους νόμους τους οποίους η ίδια προτείνει. Ευχαριστώ Ραμόν. Για τους πράσινους δεν ε, υπάρχει ομιλητής. Για την ΚΟΕ ο κύριος Βιέγκας. Δεν είναι εδώ. Ούτε άλλος κανείς ε, για τις ομάδες EFTD και η συνάδελφος Ζάνη. Πάμε στο Catch Ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση εκ μέρου του ΕΛΚ. Θέλω να πω για το άρθρο 15 ότι από τη σκοπιά του ΕΛΚ η μακροοικονομική ερεσιμότητα βρίσκεται στην καρδιά την ίδια του αμφιλεγόμενου κανονισμού. Εάν την καταργήσουμε ή την αποδυναμώσουμε, δεν μπορούμε εμεί να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε σε καμία περίπτωση, για να το πω και απλά και ξε, ξέστερα. Ähm, Ευχαριστώ πολύ ο κύριος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, άλλοι παρεμβαίνονται στο Catch the Eye. Όχι. Κανείς. Ο συνάδελφος Φέρμπερ θα κάνει μια σύνοψη. Θέλει για λογαριασμό της ε, εισηγήτριας. Ε, ευχαριστώ να συνοψίσω για λογαριασμό της Ιβάνας, αλλά ελπίζω να επικεντρωθούμε αφενός στις ε, τροπολογίες που είναι της αρμοδιότητας της ΕΚΟΝ και δεύτερον να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία να βρίσκει σύμφωνη και να ικανοποιεί την ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την υπόδειξη. Ε, και από μπάτζε, Έμπλ, Tran, Agri, Λίμπε υπάρχουν γνωμοδοτήσεις εκτός από τη δική μας. Envy, Τραν, Άγκρι, PES, Λίμπε. 20 ε, Νοεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Ωραία. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας εδώ. Πάμε τώρα στις ψηφοφορίες οι οποίες όμως ε, πρόκειτο να αρχίσουν 7 ε, και 10. 8 ε, και 10, συγγνώμη. Είναι ενδεικτικό το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα. Οπότε, καλό είναι να διακόψουμε για να έρθουν οι συνάδελφοι που έχουν λάβει υπόψη τους το ενδεικτικό πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε στις 8 και 10. So, liebe, Αγαπητοί συνάδελφοι, πήγε να πει σύντροφοι ο Πρόεδρος και διόρθωσε. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία απόψε, μία παράκληση οι συγητές και οι σκιώδεις των επόμενων σημείων να μείνουν στην αίθουσα γιατί έχουμε ένα φάκελο με πολλές συμβιβαστικές γιατί η ψηφορία θα χρειαστούμε λιγότερο από πέντε λεπτά και μετά πρέπει να ακολουθήσουμε τα θέματά μας ε, και θα τα πιάσουμε νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε το ενδεικτικό πρόγραμμα. Μην φύγετε λοιπόν. Πάμε τώρα να ψηφίσουμε σχέδιο γνωμοδότησης του συναδέλφου Φρουντσουλίκα για την μεταβλητή ολοκλήρωση. Και αρχίζομαι με δοκιμαστική ψηφοφορία. Πατήστε ένα από τα τρία κουμπάκια. Κάνουμε τεστ. Εντάξει, όλα καλά, ψήφισαν όλοι. Και οι καθυστερημένοι. Εντάξει είμαστε. Ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στην ψηφοφορία. Και πάμε κατευθείαν στην συμβιβαστική α, υπέρ. Κατά ε, δεκτή. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ε, Σ υπέρ κατά για την Σ. Α, έχουμε ε, προφορική τροπολογία. Συνάδελφο συνάδελφος Μπερές. Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά αν γίνεται θα ήθελα να κάνω πραγματική προφορική τροπολογία, προφολογία, ε, που παρουσιάζεται μόνο στην Επιτροπή. Στη συμβιβαστική ΣΥ λοιπόν, αντί να πούμε καλή την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, να πούμε καλή την θέσπιση του διαδόχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Υπάρχουν αντιρρήσεις ε, σε αυτή την ε, προφορική τροπολογία. Όχι από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, συμβαστική ΣΥ μαζί με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της ε, συμβαστικής ΣΥ μαζί με την προφορική τροπολογία. κατά αποχές ε, δεκτή. προχωρούμε στη συμβαστική D. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προχωρούμε στην παράγραφο 4, αρχικό κείμενο υπέρ κατά ε, δεκτή, παράγραφος 5 υπέρ κατά η τροπολογία 13 υπέρ κατά απερίφθη. Ε, δεν ζήτησε αποχές αλλά είναι σαφές ότι απορρίπτεται το, το πρωτότυπο, το αρχικό κείμενο. Το αρχικό κείμενο υπέρ κατά δεκτό συμβιβαστική ή υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασης ψηφοφορίας. Δεκτή. Τώρα. Πάμε στο κείμενο ως ετροποποιήθη. Υπέρ με ονομαστική, με ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ κατά αποχές. Πέρας. 31 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, μία αποχή, δεκτό το κείμενο. Ωραία. Να μείνουν οι συνάδελφοι παρακαλώ που ε, έχουν ενδιαφέρον για τα επόμενα.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 Okay, Κάποιοι που θέλετε να φύγετε, παρακαλώ να το κάνετε με ήσυχο τρόπο. Επανερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 8 είναι η ενίσχυση ε, Α, για μια στιγμή. Όχι, όχι. Προφανώς έκανα λάθος, λέει η πρόεδρος. Δεν ήθελα να πω αυτό. Μιλάμε τώρα για τους τίτλους οι οποίοι ασφαλίζονται μέσω κρατικών ομολόγων. Ο, ο Βάιτσεκερ έχει το λόγο. Γιάκομπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι βέβαιος ότι κάθε σκιώδης ε, έχει φτάσει γιατί κανονικά η συζήτηση θα ξεκινούσε στις 8.30 αλλά εν περιπτώσει. Νομίζω ότι η σημασία που έχουν αυτές οι προτάσεις σχετικά με κρατικά ομόλογα ε, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν εγγύηση στην αγορά τίτλων ε, είναι ένα σύστημα το οποίο ονομάζουμε SBs έχει τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να βρεθεί ένας καλός, ένα καλό μέσο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με το θέμα αυτό, κάτι το οποίο μέσω της νέας αυτής χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας θα την ονόμαζα, θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για το μέλλον ε, της ε, ζώνης ευρώ. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό ε, μέσω της δημιουργίας της SBBS με συμμετρικό τρόπο, δεν δίνουμε δηλαδή κάποια προτίμηση σε ένα κρατικό ομόλογο, κάτι το οποίο θα ήταν πολιτική δυσκολία αλλά και τεχνική δυσκολία γιατί προφανώς οι αξιολογήσεις δεν είναι από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης κινδύνου του διεθνούς χρηματοπιστωτικού. Έγινε λοιπόν συμμετρικό το σύστημα και αντίθετα με άλλα μέσα δημιουργής, δημιουργίας ασφαλών αγαθών ας πούμε στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη δεν απαιτούνται συγκεκριμένες εγγυήσεις. Και εδώ δεύτερος στόχος είναι να υπάρξει ε, μια δυνατότητα επιλογής από πολλούς τρόπους, ε, με πολλούς τρόπους μάλλον ε, ασφαλών τρόπων επενδύσεων, και γελάει ο Φέμπερ γιατί προφανώς ε, έχουμε από κοινού εξετάσει κάποια από τα πλεονεκτήματα και κάποια από τα μειονεκτήματα των μέσων που είχαμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας. Τρίτος στόχος και αυτός σχετικός είναι να μειώσουμε τα αποσταθεροποιητικά φαινόμενα που είδαμε στις προηγούμενες κρίσεις και που λειτουργούν αποσταθεροποιητικά ακριβώς και το θέμα είναι αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον ESM για να μην έχουμε το πρόβλημα αυτό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν προτείνει την προώθηση αυτών των μέσων. Η έκθεσή μου συγκεντρώνεται στους τέσσερις τομείς τους οποίους πιστεύω ότι υπάρχει χώρος βελτίωσης. Ο πρώτος αφορά την ρυθμιστική αντιμετώπιση των SBBS στις, στους ισολογισμούς των πιστοτικών ιδρυμάτων. Νομίζω ότι ο κανονισμός αυτός δεν θα πρέπει να έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει γενικότερα το θέμα του δημοσίου χρέους ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι δεν έχουμε ακριβώς ε, έναν κανονισμό ειδικό για όλα αυτά τα θέματα και η κατάσταση χειροτερεύει πιθανώς και δεν θα πρέπει και το SBBF να το κάνει ακόμα χειρότερο. In my report, I make a proposal... Και γι' αυτό στην έκθεσή μου κάνω μία πρόταση οποία προτείνει να έχουμε τα λεγόμενα junior tranche, mezzanine tranche και senior tranches, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων που μέχρι τώρα ε, έχουν πλέον εκτήματα και θα συνεχίσουν να τα έχουν σύμφωνα με το SBBS, αλλά αν κάποιος θέλει μόνο το κατώτερο επίπεδο, αυτό δεν θα μπορεί να το κάνει με τη δική μου τροπολογία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι μια πρώτη τεχνική λύση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Η δεύτερη πρόταση αφορά την εποπτεία. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ ήταν κάπως επιδερμική. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η αγορά θα πρέπει να είναι αγορά εμπιστοσύνης και θα ένιωθα καλύτερα αν υπάρξει ένα συγκεντρωτικό και εναρμονισμένο σύστημα πιστοποίησης από την ΕΣΜΑ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε επίπεδο μεμονωμένων εποπτικών αρχών. Και τρίτον υπάρχει το θέμα της σύνθεσης των χαρτοφυλακίων. Φυσικά και μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες αν ένα κράτος μέλος λόγω του ότι έχει ένα υψηλό πλεόνασμα θεωρεί ότι μπορεί να απαλλαγεί από ε, πάρα πολλές ή μάλλον να αγοράσει πάρα πολλά κρατικά ομόλογα οπότε τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια σπάνη των ομολόγων αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι ε, ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα και υπάρχει και πρόβλημα μερικές φορές όταν κάποιες χώρες δεν προχωρούν στην έκδοση ομολόγων τέτοιου είδους και γι' αυτό κάνουμε μία πρόταση σύμφωνα με την οποία η διαδικασία σύνθεσης του χαρτοφυλακίου μπορεί να τροπολογηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε οι εκδόσεις SBBS να μην παγώσουν κατά κάποιο τρόπο από τις καταστάσεις τις οποίες προανέφερα. Αυτό δεν το επέτρεπε η Επιτροπή στην αρχική πρόταση και υπάρχει και ένα επιπλέον σημείο που λέει ότι το θέμα της αναδιάφρωσης και εδώ οφείλω να αποδώσω ε, ε, τιμή σε σχέση με την έκθεση που κυκλοφόρησε για τα SBs. Υπάρχει ένα κεφάλαιο για τον τρόπο αντιμετώπισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στην περίπτωση αναδιάφρασης του χρέους μιας χώρας μέλους όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν συμπτώσεις συμφερόντων ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα, το senior, mezzanine και junior. Και γι' αυτό ακριβώς καταθέσαμε αρκετές τροπολογίες προσπαθώντας να βρούμε κάποιες ε, α, λύσεις οι οποίες να είναι προληπτικού τύπου και τις οποίες μπορεί να ελέγχει το ESM. Συνεπώς λοιπόν η πρόταση SBBS βασίζεται σε μια εξαιρετική ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να είναι ένας βασικός τρόπος για την πορεία μας τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, το πρόβλημα της απουσίας μιας ασφαλούς δυνατότητας στον τομέα των επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης υπάρχει και το θέμα εδώ ε, της προετοιμασίας του επόμενου βήματος ε, ο κανονισμός αυτό προσπαθεί νομίζω να το κάνει και μπορεί να το πετύχει και ε, εγώ ευχαριστώ ε, για τις τροπολογίες των σκιωδών είχαμε καλές συναντήσεις μαζί τους και ελπίζω να συνεχιστεί η συζήτηση Ευχαριστώ Ιάκωβ. Εάν Κάποιοι από τους βοηθούς ε, στην αίθουσα ξέρουν ότι συζητιέται το θέμα αυτό. Εδοποιήστε όποιον είναι αρμόδιος να έρθει όσο γίνεται το πιο γρήγορα, γιατί θα περάσουμε από το ένα σημείο της ημερήσιας στο άλλο. <clears throat> Τηλεφωνήστε τους για να έρθουν, διότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ακριβώς το πρόγραμμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Είναι ενδεικτικό. Θα προχωρούμε λοιπόν ώστε να είναι πιο γρήγορο. Τηλεφωνήστε τους και τώρα να ζητήσω από τους Χιώδης να κάνουν τα σχόλιά τους. Η κυρία Χούμπνερ. Ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ τον Γιάκο Μπρένερ τόσο ενθουσιώδης για πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά θα πρέπει να ε, σας διαβάσω το σχολείο της αδέλφου που είναι γεμάτο ενθουσιασμό για εσά, Γιάκομπ. Είναι χαρά μου λοιπόν πολλέ ευχαριστίε στην συνάδελφο Ντανούτα που με εκπροσωπεί σήμερα. Ε, με συγχωρείτε που δεν μπορούσα να είμαι εδώ η ίδια. Ε, εργαζόμαστε επί του θέματο αυτού, εξώγραφου που υποστηρίζονται από κρατικά ομάλογα, και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε δυναμίε και ελλείψει στο συγκεκριμένο τομέα. Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι το θέμα αυτό με τον κύριο Γιάκομπ Φων και τον σκιώδη συγκεκριτή για το θέμα αυτό και ήταν μια πολύ οικοδομητική ε, εργασία σε συνεργασία με του υπόλοιπου σκιώδη. Εδώ και εβδομάδε έχουμε τονίσει διαφορετικέ πτυχέ που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και συμφωνώ απολύτω με του στόχου τη πρόταση, ε, την ε, μείωση του κινδύνου ω ένα κλειδί για την επιτυχία σταθερή σταθερότητα. Ε, την επίτευξη μάλλον σταθερότητα. Θα πρέπει να περιορίσουμε το συσχετισμό μεταξύ των κρατικών ομολόγων και το τραπεζικό τομέα όμω. Και θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση ε, με τι τροπολογίε που θα υποβληθούν σχετικά. Η ευνοϊκή ε, μεταχείριση των branches είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε θετική συνεννόηση και και θετικό συνδυασμό των διαφόρων προτεραιοτήτων, αλλά με σκοπό να εξυπηρετήσουμε την Ευρώπη μας. Ευχαριστώ πολύ. Συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Φων Βάιτσεκερ για την ωραία έκθεση, ιδιαίτερα το ανοιχτό κλίμα συζήτησης και με τα πάνελ εμπειρογνωμόνων που κάνατε. Είμαι λιγότερο ενθουσιώδης από εσά σε σχέση με αυτή την πρόταση, το ξέρετε θα παρουσιάσω κάποιες επιφυλάξεις. Το πρώτο θέμα είναι αν για το προϊόν αυτό υπάρχει κατάλληλη αγορά ή ανάλογη αγορά. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Υπάρχει και στη μελέτη επιπτώσεων και στις μελέτες της Κομισιόν. Ήταν ένα θέμα πάντα αυτό. Πρώτα θα αναπτυχθεί η αγορά όταν το ρυθμιστικό προνόμιο μειωθεί και απαλληφθεί. Και εδώ σε ένα κρίσιμο θέμα στην έκθεση, γιατί η πρότασή σας ε, να έχουμε πλήρη ρυθμιστική ε, πλήρες ρυθμιστικό προνόμιο ακόμα και όταν τα SBBS ε, είναι σωστά κατανεμημένα ανάμεσα σε τμήματα ίσονος μέσης ανώτερης εξασφάλισης εκεί είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα γίνει και θα είναι δύσκολο να ε, ε, ε, δυσκολέψουμε την αγορά κρατικών ομολόγων ε, περιλαμβάνοντας ένα νέο τύπο, ένα νέο είδος, εισάγοντας το θετικό ρίσκο για τα κρατικά ομόλογα θα πρέπει να ε, συμπεράνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει στάθμιση κινδύνου και για άλλους τίτλους. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό το σύστημα ανταποκρίνεται στην γενικότερη λογική που είχατε παρουσιάσει. Το δεύτερο σημείο που δεν μου αρέσει στην πρόταση της Κομισιόν είναι αυτή η συμμετρία που εσείς την επενέσατε γιατί δεν έχω πιστεί, για να σας το πω έτσι, ότι θα πρέπει να είναι τόσο υπερβολική η ρύθμιση όπως προβλέπετε. Να προδιαγράψουμε δηλαδή ότι οι κρατικοί τίτλοι, τα κρατικά ομόλογα θα ε, τηρούνται ε, αναλογικά στα διάφορα τμήματα. Καλύτερα να αναλάβει η αγορά την εξασφάλιση των ε, κρατικών ομολόγων ε, με μορφή διαφορών τίτλων και να χωρίσουν εκείνη στα τμήματα Νομίζω ότι θα ήταν μεγαλύτερη η ασφάλεια από ό,τι προβλέπει το σύστημα με τα SBBS. Η ασφάλεια των SBBS, ακόμα και με την ε, πρόβλεψη των τμήματων αμφισβητείται γιατί υπάρχουν κίνδυνοι ε, σε 19 κράτη της Ευρωζώνης ε, υπάρχουν προβλήματα με τα κρατικά ομόλογα και αν υπάρχει ε, κάποια πτώχευση μπορεί να υπάρχουν ε, ε, αρνητικά αποτελέσματα και επιπτώσεις και σε άλλους. Και δεν νομίζω ότι το Τμήμα Ανώτερης Εξασφάλισης καλύπτει επαρκώς το θέμα. Δεν πρέπει να προδιαγράψουμε αναλογικότητα σε σχέση με τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων οριζόντια στα κράτη της Ευρωζώνης. Μπορεί να επιτρέπουμε να ε, αποφασίσει η αγορά για το μέγεθος αυτού του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης το 17% έχει αμφισβητηθεί αν είναι αρκετό. Και υπάρχει και ένα σενάριο που δεν το θεωρώ το πιο λογικό φανές, ε, δηλαδή η πτώχευση της ε, Γερμανίας, αλλά ε, δεν ξέρουμε αν το 70% ε, είναι αρκετά ασφαλές και μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν μικρότερα ε, τμήματα ανώτερης εξασφάλισης και τα υπόλοιπα να περάσουν στο μέσο ή το ίσονος εξασφάλισης τμήμα. 5%. Εγώ είχα προτείνει 10%. Αλλά αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και να δούμε τι, λένε, τι λέει η πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ε, εκ μέρους της άλλης, το κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό Είναι ιδιαίτερα ευρωπαϊκός αυτός ο ενθουσιασμός. Η πρόταση είναι πολύ καλή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς μπορεί να βελτιωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγχαίρω για την προσπάθεια την οποία έκανε ο εισηγητής ε, και η σωστή προετοιμασία μέσω της επαφής με τους εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί Τώρα δεν θα εμπλακώ εγώ σε τεχνικές λεπτομέρειες γιατί πάντα θα υπάρχουν ε, αμφιβολίες σε τεχνικό επίπεδο για λεπτομέρειες αν θα είναι 70% ή 75%. Αυτό που έχει σημασία είναι η πολιτική βούληση. Υπάρχουν κάποιες ιδέες. Εμείς φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες δεσμεύσεις ε, για τις τράπεζες σε σχέση με τις χώρες προέλευσης αν έχουμε σαν στόχο να δημιουργήσουμε μία ισχυρή εσωτερική αγορά θα πρέπει να μην είναι απόλυτα δεσμευμένες με το δημόσιο χρέος της χώρας τους οι τα πιστοτικά ιδρύματα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε λοιπόν την δυνατότητα ανάκαμψης του συστήματος και τις οικονομικές δυνατότητες γενικότερα είναι σαφές ότι η εκδότρια αρχή θα πρέπει να, έχει, ε, να είναι ειδικού στόχου. Δεν θα πρέπει δηλαδή να αναπτύσσει διαφορετικές ε, δραστηριότητες. Πρέπει να είναι ένα SPE. Ε, και το βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης αρχής, του συγκεκριμένου μέσου, είναι ότι είναι ευρωπαϊκό. Είναι σημαντικό επίσης να δούμε ακριβώς και τι γίνεται με τη ζήτηση ε, χαμηλού κινδύνου τίτλων σε ευρώ και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακριβώς την κάλυψη αυτών. Είναι λοιπόν επίσης πάρα πολύ σημαντικό και πέρα από αυτά τα οποία είπαμε ε, για τις εκδότριες αρχές ε, και να υπάρχει μια σωστή εποπτεία των εκδοτών, των SBBS, που θα πρέπει να καλύπτονται από την ΕΣΜΑ. ΕΣΜΑ λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, νομίζω ότι αυτό είναι που ολοκληρώνει αν θέλετε τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών αυτών των τίτλων. Νομίζω ότι πρόκειται για, ένα, για πλήρη περίπλοκα μέσα και τίτλους, αλλά είναι κάτι το οποίο καλύπτει τις ανάγκες και των εκδοτών και των καταναλωτών. Τώρα σχετικά με το κατώτερο επίπεδο, ε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε μεμονωμένους καταναλωτές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε μία λύση ε, με ενθουσιασμό. Έχω τώρα και κάποιες άλλες αμφιβολίες, αμφιβολίες συγγνώμη, σε σχέση με τη συμπεριφορά των μέσων αυτών σε περιπτώσεις κρίσης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε θετικοί απέναντι στην πρόταση αυτή για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ε, ε, ε πρέπει να λειτουργήσουμε σε πολιτικό επίπεδο και έχουμε δύο ε, απόψεις για την Ευρώπη μπροστά μας. Έχουμε εδώ μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στο μέγιστο βαθμό. Και το είπε και ο κύριος Βαϊτσέκερ. Δεν θα πρέπει να το ονοματίζουμε, να το αποδίδουμε διαφορετικά. Νομίζω ότι δεν είναι υποκατάστατο των ευρωομολόγων. Σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο τα ευρωομόλογα μπορεί να είναι κάτι το απαραίτητο. Για τους πρασίνους... Ο κύριο Ουρτασούν, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και για την εξαιρετική προετοιμασία του όλου φακέλου. Πραγματικά ε, κάναμε πολλέ ενδιαφέρουσε ακροάσει με τη συμμετοχή πολλών ειδοπυρογνωμόνων που είχαν ε, επικοδομητική συνεισφορά στη δουλειά μα. Το πρώτο που θέλω να πω, το είπατε και εσεί στι αγωγικέ σα παρατηρήσει και στη δήλωσή σα, είναι το εξή. Προσπαθούμε να βρούμε μία ιδανική λύση σε κάτι που έχει να κάνει όμως με την ε, μεταρρύθμιση την διορθωτική. Αυτό είναι και η ουσία της συζήτησης. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε εδώ τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία του ενεργητικού ή τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Αυτό πρέπει να είναι λοιπόν ευθύ εξ αρχή ξεκάθαρο στα μυαλά όλων όταν σκέφτονται αυτό το θέμα. Επίση, ε, σε σχέση με τι προτάσει που υποβάλαμε, και τις έχει εξετάσει ευνοϊκά ο εισηγητής, τις ανέφερε, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για τον αρνητικό αντίκτυπο ως προς την κρίση και τις επιπτώσεις της. Τα είδαμε αυτά σε κάποιες από τις ακροάσεις, τα συζητήσαμε και επίσης ο εισηγητής ανέφερε ότι τα SBS, SBBS δεν ε, σχετίζονται σωστά με το τραπεζικό σύστημα το πρόβλημα της ασφάλειας από τα ε, ομόλογα αυτά είναι θέμα των εγγύσεων. Και για τις μικρότερες χώρες ξέρουμε ότι οι ερνητικές συνέπειες είναι περισσότερες ε, και πιο πιθανές για αυτές. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται με τα ομόλογα που αναφέρει στην πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το crying out κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ε, ρευστότητα των δηλαδή, μελών. Καθώ δημιουργούνται αυτά τα ομόλογα. Τώρα, σε σχέση με τι συγκεκριμένε προτάσει του εισηγητή, καλωσορίζω κάποια από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν. Και κατά πρώτον, συμφωνούμε ότι η ρυθμιστική μεταχείριση των SPBS, ε, των junior, θα πρέπει να αλλάξει ε, από τις τράπεζες ιδίω και το ίδιο και το σύστημα εποπτείας. Κάτι που κατάλαβα ότι και εσείς επιθυμείτε με την παρέμβασή σας. Επίσης πρέπει να έχουμε κάποια εχέγγυα για να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις ε, στην αγορά κρατικών ομολόγων εφόσον εκδοθούν τέτοιου είδους ομόλογα, αξιόγραφα και να δούμε τι προϋποθέσεις χρειάζονται ένα ακόμη σημείο είναι ότι θα πρέπει να υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον. Προτού πληγούν αρνητικά λοιπόν οι διάφοροι μέτοχοι, οι κάτοχοι των ομολόγων, θα πρέπει να δούμε την αρνητική, τις αρνητικές επιπτώσεις του εργαλείου και να τις μελετήσουμε σενάρια. Συνολικά λοιπόν, να πω ότι παρόλο που κάπως επιφυλακτικοί είμαστε για το ρόλο των SBBS, Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι λύση βεβαίω για τα πραγματικά στοιχεία ενεργετικού, αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να έχουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν εδώ από την ΚΟΕ ή από την EFTD, αλλά θα ζητήσω τον κύριο Τζάνι να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί τα πιο σημαντικά νομίζω ήδη ακούστηκαν από τους προηγούμενους συναδέλφους. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρότασή του. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να προωθηθεί αν και υπάρχουν κάποια από τα προβλήματα τα οποία ήδη συζητήσαμε στην πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι το set allocation της πρότασης ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που πρέπει να επανεξεταστεί. Το θέμα της ε, διαφάνειας πρέπει να επανεξεταστεί, της πιστοποίησης. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτοπιστοποίηση, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας πραγματικός έλεγχος από πλευράς των αρμοδίων εποπτικών αρχών. Είμαι ιδιαίτερα διστακτικός σε σχέση με το σύνολο της πρότασης έχει πολλά αρνητικά σημεία. Νομίζω ότι ο Γερμανός συνάδελφος πριν από μένα αναφέρθηκε στις δυνατότητες της αγοράς να απορροφήσει αυτού του τύπου τα μέσα και την αποτελεσματικότητα του μέσου αυτού να δημιουργήσει ελεύθερα κινδύνου μέσα και έρχομαι σε αυτό που είπε και ο Ούρτασον εδώ για μια ακόμη φορά δηλαδή τα ευρωπαϊκά όργανα μπροστά από την δυσκολία τροποποίησης και αλλαγής ε, της δυσλειτουργίας που τα χαρακτηρίζει σε ορισμένους τομείς, αναζητούν να βρουνε μια λύση η οποία να είναι φιλόδοξη, περίπλοκη, να περιλαμβάνει και μια μηχανική σε εισαγωγικά χρηματοπιστωτική και ακριβώς ε, λόγω του ότι είναι εσκεμμένος ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωζώνης ως ε, χώρου ε, χωρίς απουσία κινδύνου σε σχέση με, τις, με τους τίτλους τους διαθέσιμους και τα ομόλογα είναι δύσκολο να ξεφύγει κανείς από μια αντικειμενική δυσκολία όσο περίπλοκες και να είναι οι ρυθμίσεις. Δεν είναι δυνατόν να βρούμε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι απαλλαγμένο από κάθε τύπο κινδύνου. Νομίζω ότι το μέσο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους τους οποίους ήδη αναφέραμε αλλά να είναι και κάτι το ενδιαφέρον για τους ε, ιδιώτες ε, καταναλωτές που θα πρέπει να ενδιαφερθούν για αυτού του είδους ε, τους τίτλους. Λοιπόν, catch the eye, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να θέσει κάποιες ερωτήσεις. Όχι, φαίνεται ότι θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Φον Βάιτσέκερ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι διότι η ατμόσφαιρα της συζήτησης απόψε επιτρέπει, παρά τις διαφορές που σαφώς υπάρχουν κάποιες, να γίνει πολύ ουσιαστική συζήτηση. Λοιπόν, να επικεντρωθώ σε κάποιους τομείς που νομίζω είναι σημαντικοί. Το πρώτο είναι ένα θέμα στρατηγικής. Και αυτό αναφέρεται σε αυτό που είπε και ο Μπερντούκας και αυτό που είπατε και εσείς. Πρόκειται για το πόσο μπορούμε να λύσουμε, πόσα μπορούμε να λύσουμε σε αυτό το στάδιο με αυτό το φάκελο. Για παράδειγμα, συμφωνώ ε, θεωρητικά μαζί σας ότι για να ολοκληρωθεί η εικόνα Χρειάζεται μία πλήρης λύση στο πρόβλημα του δεσμού τραπεζών κρατών και κυβερνήσεων. Ε, αυτό θα απαιτούσε κάποιο δούνε και λαβίν ε, από... μεταξύ χωρών που είναι σταθερές και άλλες που ακόμα παλεύουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε ε, ένα άλμα ή να καταπιούμε μια μπουκιά πολύ μεγάλη για αυτό που δυνάμεθα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ένα πρώτο βήμα χωρίς να το μετανιώσουμε. Συμφωνούμε ότι ε, τώρα η αγορά δεν είναι τεράστια. Η αγορά θα αναπτυχθεί όταν υπάρχει ένα ε, προνόμιο στο τμήμα ε, ίσονος εξασφάλισης ε, που δεν θα ε, κάλυπτε όλους τους ε, τίτλους. Αν δημιουργηθεί όμως θα διευκολύνει τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις για να γίνει ε, μια συμφωνία πακέτο που θα περιλαμβάνει και τα SBBS. Έτσι θα είναι πιο σταθερό το νόμισμα στην Ένωση και θα ε, είναι και τα κίνητρα λογικά σε αυτή την ε, ένωση. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Γι' αυτό ε, επικεντρώνουμε στο τμήμα ίσονος εξασφάλισης που πρέπει όμως να προσεχτεί για να μην ενισχυθεί περισσότερο δεσμός κράτους τράπεζας. Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Είναι ένα πρόβλημα καθ' αυτό που θα πρέπει να το δούμε ε, από μόνο του στο επόμενο βήμα. Αλλά δεν θέλω η πρόταση για τα SBBS να χειροτερέψει τα πράγματα εκεί. Οπότε θα, μια προσέγγιση που είναι προσεκτική για να μην μετανιώσουμε, δεν είναι μεγάλη επίβολη που ισχυρίζεται ότι θα λύσει όλα μας τα προβλήματα. Το πρόβλημα της ρευστότητα που είπατε κι εσείς εδώ πραγματικά πρόκειται για μια συναλλαγή και βεβαίως όλα έχουν ένα κόστος. Αυτό μην το ξεχνάμε. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα. Πώς θα γίνει. Θα βάλουμε τα SBBS μέσα σε ένα, μια συμφωνία πακέτο μαζί με μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, ε, μηχανισμούς αντιμετώπισης διαρροής κεφαλαίων, ε, ε, τα τμήματα μπορεί να βοηθήσουν εδώ και μπορεί να γίνει και προληπτικός δανεισμός που θα διευκολύνεται έτσι και θα υπάρχει και το ECB. Και σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, αν η αλληλεπίδραση είναι καλά σχεδιασμένη μεταξύ αυτών των μηχανισμών, κατά πάσα πιθανότητα θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Αλλά και πάλι, απομονωμένα δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Δεν πειράζει όμως, γιατί ε, απομονωμένη η αγορά των SBBS, η αγορά θα είναι μικρή ούτως ή άλλως. Εγώ ως εκεί πάω σήμερα, περιμένω με ενδιαφέρον τις επόμενες συναντήσεις των σκιωδών που έχουν ήδη προγραμματιστεί και περιμένω και τις εκθέσεις σας και θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα σε αυτό το θεματολόγιο, αλλά λιγάκι να πάμε πιο μπροστά όλοι μαζί και με τη βοήθεια του ΕΛΚ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων ε, για την παρέμβαση της Ντανούτα και με τον ε, συνάδελφο Μαρτιτσέλη ήταν πολύ επικοδομητικές οι συζητήσεις για να προχωρήσει ο φάκελος, να προχωρήσουν τα θέματα. Και στο Συμβούλιο υπάρχουν και κάποια ε, προβλήματα, ανασταλτικοί παράγοντες. Μπορεί να μην ξεπεράσω με τον μπλοκάρισμα που υπάρχει, μπορεί να μην προλάβουμε σε αυτή τη θητεία. Αλλά αν έχουμε μια στέρεη θέση ως Κοινοβούλιο, αυτό βοηθάει και τη σκέψη του Κοινοβουλίου. Μπορεί να βοηθήσουμε να ξεπεράσει και το Συμβούλιο τις δυσκολίε που έχει. Ε, αυτό πρέπει να στοχεύσουμε. Ευχαριστώ κύριε Φων Βάιτσέκερ. Ε, θα σας δώσω το χρονοδιάγραμμα. Ε, στις 20 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και η εξέταση στις 10 Δεκεμβρίου των τροπολογιών και η ψηφοφορία αρχές του Ιανουαρίου του 2019. Ψηφοφορία στην ΕΚΟ. Ε, αυτά ελπίζω να είναι αποδεκτές ε, ε, ημερομηνίες. Χωρίς διάλειμμα πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ήρθε η συγγήτρια είναι εδώ. Το επόμενο είναι η ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και του μεσοπρόθεσμου με δημοσιονομικού προσανατολισμού στα κράτη-μέλη. Δίνω καταρχήν στην κυρία Χιούμπνερ το λόγο για να μας πει τις παρατηρήσεις Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτό είναι άλλο θέμα εδώ έχουμε μεγάλη διέρεση και στην Επιτροπή και μάλλον και στο Κοινοβούλιο και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Πρόκειται για τη μεταφορά στην εσωτερική, στην εθνική νομοθεσία του μεγαλύτερου μέρους του άρθρου 3 ε, τη συνθήκη για τη σταθερότητα, συντονισμό και διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ε, πήρα πολλές προτάσεις. Ε, αρκετές ομάδες οι σοσιαλιστές, οι γκουε, οι FDD και οι πράσινοι ζητούν την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν μέσα από τις τροπολογίες τους. Και πρέπει να πω ότι με δυσκολεύει αυτή η προσέγγιση. Δεν τίνω να στηρίξω μια τέτοια προσέγγιση Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, αυτό το κομμάτι δηλαδή ε, της ε, δημοσιονομικής συνθήκης. Επίσης, αν απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν, αυτό θα ήταν πολύ αντιπαραγωγικό, ακόμα και για εκείνους που δεν συμφωνούν με το τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, από πολιτικής πλευράς θα ήταν ε, επιβλαβές για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρόκειται για μια διαδικασία διαβουλεύσεων. Το Συμβούλιο πρέπει να πάρει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά η θέση αυτή δεν είναι δεσμευτική κατ' ουδένα τρόπο για το Συμβούλιο. Αν συμφωνήσουμε να απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν, αυτό δεν θα σταματήσει τις διαδικασίες στο Συμβούλιο. Επίσης, θεωρητικά, αν το Συμβούλιο το ίδιο απορρίψει την πρόταση, αυτό δεν θα σήμαινε ότι κάποιο στοιχείο του τωρινού δημοσιονομικού πλαισίου θα καταργεί το. λεγόμενο εξάπτυχο, το δίπτυχο θα εξακολουθούσαν να ισχύουν όπως έχουν. Η απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν θα ήταν μια πολιτική δήλωση, αναμφιβόλως, αλλά νομίζω ότι θα αποστείλουμε μηνύματα που δεν είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα, να στείλουμε το μήνυμα ότι δεχόμαστε τις διακυβερνητικές λύσεις, ότι δεν έχουμε πρόβλημα με αυτές. Αυτό θα σήμαινε ότι θα ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη θέση μας, ίσως θα θυμάστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη μάχη για να συμπεριληφθούν ε, να, να, συμπεριληφθεί στην θήκη το άρθρο 16 που υποχρεώνει την ε, ε, τήρηση της συνθήκης. Θα θυμάστε ότι αυτό αντιβαίνει σε προηγούμενες θέσεις του Κοινοβουλίου από το 2015 η έκθεση για την, ε, την επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου. Είπαμε ότι η δημοσιονομική συνθήκη που είναι εκτός των δομών των θεσμικών οργάνων της Ένωσης είναι ένα βήμα πίσω για την πολιτική ολοκλήρωση και είχαμε ζητήσει τότε πλήρη ολοκλήρωση στο κοινοτικό πλαίσιο το 2017 επίσης ε, επίσης ε, εγκρίναμε μια έκθεση όπου αναφερόταν αυτό το θέμα ως απέτηση του Κοινοβουλίου και σε όλες τις εκθέσεις για την Τραπεζική Ένωση τα σώμεθα κατά της διακυβερνητικής συμφωνίας που ζητεί την ενσωμάτωση άλλων διεθνών ε, μέσων. Νομίζω και ελπίζω ε, και, θεωρώ ότι εμείς ως Κοινοβούλιο όταν απορρίψαμε τις ε, διακυβερνητικές λύσεις είχαμε κάποιους λόγους γι' αυτό. Και το δεύτερο θέμα που ήθελα να αναφέρω, έχοντας διαβάσει τις τροπολογίες σας, είναι ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για μεταφορά στην εσωτερική νομοθεσία αυτού του, του, του τμήματος της συνθήκης, θα μας ε, ε, κάνει να χάσουμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου στις περαιτέρω συζητήσεις και επανεξετάσεις του δημοσιονομικού πλαισίου. Με την προτινόμενη οδηγία νομίζω ε, και σχετικά με τις διατάξεις της δημοσιονομικής συνθήκης περνάμε σε διαφορετικό νομικό καθεστώς. Το Κοινοβούλιο παλιότερα δεν είχε κανένα ρόλο, σε, καμία φάση σχετικά με το νομικό, σχετικά με το νομικό καθεστώς υπό το οποίο θα ε, γίνονταν διαβουλεύσεις με το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκείνο το τελευταίο θα μπορούσε να, δώσει, να γνωμοδοτήσει. Γιατί να μην ε, χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται να αποκτήσουμε μεγαλύτερη επιρροή στη δημοσιονομική πολιτική. Υπάρχουν διάφορες γνώμες, και κυρίως από το Άλντι και την, ε, και την ομάδα ECR, που προτείνουν προσαρμογές στο κείμενο της Κομισιόν και υπάρχουν και άλλες απόψεις που είτε απορρίπτουν, οι πράσινοι εκτός από την απόρριψη προτείνουν και κάποιες πολύ βαθιές ουσιαστικές αλλαγές στην οδηγία. Να πω λοιπόν ότι αν συμπεριλάβουμε διατάξεις στην οδηγία αυτή που είναι αντιφατικές προς το εξάπτυχο και το δίπτυχο και την ίδια τη δημοσιονομική συνθήκη, διατρέχουμε τον κίνδυνο σύγκρουσης νόμων και εφαρμογής των νόμων, γιατί θα υπάρχουν πολλά στοιχεία στην κοινοτική νομοθεσία επί του ιδίου θέματος που θα υπαγορεύουν όμως διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και αυτό δημιουργεί νομική ανασφάλεια και μεγάλη περιπλοκότητα σε πολύ σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η πιο λογική στρατηγική και που την προτείνω είναι να γίνει η μεταφορά με τρόπο που δεν θα είναι διαταρακτικός, που θα είναι ουδέτερος σε σχέση με τις εθνικές επιλογές που έχουν γίνει για την μεταφορά στην Εθνική Νομοθεσία της Συνθήκης και νομίζω και, και ε, ε το δημοσιονομικό έλεγχο. Νομίζω ότι ε, βλέπουμε ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου ε, αρχίζει. Είμαστε τώρα στο, στην ε, προκαταρκτική διαδικασία και θα εξεταστούν το 2019 και αυτά τα νομοθετικά μέτρα, οι δέσμες νομοθετικών μέτρων που λέγονται εξάπτυχο και δίπτυχο. Και νομίζω ότι και τα δύο, αυτά οι δύο δέσμες και, το, και το δίπτυχο και τρία τέταρτο εξάπτυχου ε, αλληλο, είναι αλληλένδετες. Αν συνεχίσουμε ε, αυτή τη διαδικασία του χρόνου θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Νομίζω ότι αν καταργήσουμε τις διακυβερνητικές λύσεις και ε, τις απορρίψουμε δεν θα ε, Λύσω με κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. αλλά ήμουν άρρωστη όταν ε, παρουσιάστηκε η έκθεση και ήθελα να έχω μια ευκαιρία να πω και εγώ τις απόψεις μου. Ευχαριστούμε κυρία Χούμπνερ, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεδομένως Νομίζω ότι εδώ έχουμε πολύ σημαντικές πολιτικές διαφορές. Για μας τους σοσιαλιστές το θέμα δεν είναι ένα θεσμικό θέμα. Σε επίπεδο θεσμικό, σε καθημερινή βάση κάνουμε πράγματα και τα ξεκάνουμε επίσης εύκολα. Το θέμα είναι να δώσουμε ένα μήνυμα προς συμφέρον του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Μετά από την οικονομική κρίση του 2008, αποφασίστηκε να ληφθούν δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία ήταν μάλλον απαραίτητα. Τα μέτρα αυτά, τα οποία είχαν σαν στόχο τη σωστή εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών και ένα ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο, οδήγησαν δυστυχώς στην αποκλιμάκωση των οικονομικών δικτών των τελευταίων χρόνων, δημιούργησε προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες, στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς δεν είμαστε υπέρ της συμπερίληψης του πακέτου αυτού στις συνθήκες αν δεν υπάρξει μια σοβαρή αξιολόγηση και μια σε βάθος ε, ε, αλλαγή του πακέτου αυτού. Νομίζω ότι το σύμφωνο αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα άλλο σύμφωνο το οποίο να προσθέτει στον τομέα σύγκλησης ε, όχι αποκλειστικά αναλύοντας ε, τα δημοσιονομικά στοιχεία χωρίς ένα ευρύτερο ε, πλαίσιο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς και οικονομικούς δείκτες και όχι μόνο δημοσιονομικούς. Υπάρχουν άλλες λύσεις, έχουμε το πορτογαλικό παράδειγμα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γι' αυτό εμείς έχουμε καταθέσει μία τροπολογία απόρριψης της πρότασης σχετικά με το σύμφωνο. Δεν υπάρχει λόγος να το συμπεριλάβουμε στη συνθήκη έτσι ως έχει σήμερα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι που είναι σύντομη και περιεκτική η έκθεση της εισηγητρίας το ίδιο θα ήθελα να ακούσω και για την ε, ουσία των τροπολογιών. Υπάρχουν κάποιε τροπολογίε όμω που προτείνουν την απόρριψη τη πρόταση τη Επιτροπή ε, Σιλίβδιν. Και αυτό κάπω με οδηγεί σε σύγχυση. Διότι ξέρω πόσο δύσκολο είναι τη χώρα μου να ξεφύγει από την οικονομική κρίση και το θυμάστε όταν συζητήσαμε και το θέμα τη διακυβερνητική συνθήκη και το δημοσιονομικό σύμφωνο. Καταλαβαίνετε ότι στου συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ έχουμε αντιπροσωπείε που δεν συνυπέγραψαν τη συνθήκη και μείναν εκτός συμφώνου. Ταυτόχρονα όμως να θυμίσω ότι το σύμφωνο μάλλον η συνθήκη σταθερότητας και διακυβέρνησης της ε, οικονομικής διακυβέρνησης έχει ήδη συναυτεί από το 2012 και από, τους 25, από τα 25 συμβαλόμενα μέρη της TSG ε, οι περισσότεροι είναι και συμβαλόμενα μέρη του Δημοσιονομικού Συμφώνου και συμφωνούν ότι μέσα σε πέντε χρόνια ε, από τότε θα έπρεπε να έχει αυτό συμπεριληφθεί στο κοινοτικό δίκαιο, στο ενωσιακό δίκαιο. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα μερικά μέρη της, μέλη της Επιτροπής μας βλέπουν ε, ως ε, ανεπιθύμητη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι απλώς χρειάζονται βελτίωσεις, αλλά και οι κοινώς συμφωνημένοι κανόνες πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Υπάρχουν όρια στην ευελιξία ε, και το τι θα πρέπει να γίνει με τις επενδύσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όμως κάποια κρατημέλη είδαμε ότι κατάφεραν να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση παραμένοντας πιστά στους κανόνες του οικονομικού συμφώνου, του δημοσιονομικού συμφώνου παρά παραβιάζοντάς τους. Υπάρχει και κάτι που ονομάζεται ανεξάρτητη φορεί. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτοί οι ανεξάρτητοι φορεί όντω δεν επηρεάζονται από κανέναν, ότι δεν έχουν ευθύνε για τη χάραξη πολιτική και ότι δεν αποφαίνονται για θέματα που ξεπερνούν τα όρια των αρμοδιοτήτων του. Παρομοίω, τα μέλη του πρέπει να διορίζονται όχι μόνο βάσει τη εμπειρία του, αλλά και βάσει των προσόντων του και τη ε, ασχέτω τη πολιτική του προσχώρηση. Γι' αυτό λοιπόν εν γέννη ε, καλωσορίζω τι τροπολογίε και των υπόλοιπων μελών τη Επιτροπή μα και αναμένω τις ε, συζητήσεις που θα έχουμε για το θέμα αυτό, τις οποίες ελπίζω να είναι καρποφόρες. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω κανέναν εδώ από την Άλντε για το θέμα αυτό, οπότε τώρα να πάμε στους πρασίνους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα σφάλματα είναι ανθρώπινα, αλλά το να επιμένει κανείς είναι κάτι που είναι διαβολικό. Εράρε humanum, perseverare diabolicum. Λατινικά. Σας άκουσα με προσοχή. Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω για αυτό που λέτε. Μα θυμίζετε διαρκώ ότι έχουμε πολλά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που λένε ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο θα πρέπει να γίνει μέρος του ενουσιακού δικαίου. Να είμαστε εδώ συνεπείς και να θυμόμαστε ότι στο σε όλα αυτά τα ψηφίσματα αμέσως μετά λέγεται μετά από αξιολόγηση και αναθεώρηση αυτό δεν συμβαίνει. Κανένα, τέλο πάντων όχι κανένα, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν αμφισβητεί την ουσία τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Και να το πω ξεκάθαρα. Δεν μπορούμε ότι μπορούμε να έχουμε νομισματική ένωση χωρίς κοινού κανόνε. Παρομοίως όμως δεν μπορούμε να έχουμε και νομισματική ένωση χωρί ισχυρή και όταν λέω ισχυρή εννοώ άλλα γερμανικά, ε, ισχυρή, ε, ισχυρό μηχανισμό αλληλεγγύη. Βλέπω εδώ μια πλειοψηφία που μπορεί, κάπως νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει νομισματική ένωση με κοινό ε, νόμισμα, κοινή κεντρική τράπεζα, κοινού κανόνες και φτάνει. Δεν είναι έτσι. Ε, έχουμε υποβάλει λοιπόν τροπολογίες για την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπή και όχι γιατί δεν θέλουμε ε, νέους κανόνες, αλλά γιατί, και το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, γιατί οι κανόνε που τώρα ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων και των συνθηκών, δεν έχουν κανένα επιστημονικό έρισμα. Το 3%, το 60% είναι εντελώς πολιτικού χαρακτήρα αριθμοί. Δεν έχουν κανένα ε, επιστημονικό έρισμα. Είμαι μηχανικός. Ξέρω ότι με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι εάν λαμβάνουμε αποφάσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Έχω ακούσει πολλά ε, ψευδεπιστημονικά στοιχεία για να υποστηριχθούν ε, κάποιες θεωρίες. Οι επιστήμονες μας δίνουν και πολλές ε, ενδιαφέρουσες πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε δημοσιονομικούς κανόνες που δεν βασίζονται σε τίποτε το επιστημονικό και μάλιστα έχουν αποδείξει ότι ε, δεν αντιστέκονται στις αλλαγές των οικονομικών κύκλων. Είναι υπέρ, ε, τους καλλιεργούν τους κύκλους της οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν να τους διορθώσουμε και να τους αλλάξουμε, όχι για να τους πετάξουμε στον καλάθο των αχρήστων, να τους αναθεωρήσουμε, να γίνουν κάτι που οικονομικά να έχει νόημα, να λαμβάνουν επίσης υπόψη αυτό που είπε κάποιος, ότι οι κανόνες πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κόσμου δεν μπορεί να δεχτώ ότι οι χρηματαγορέ είναι εκπρόσωπο του λαού, του κόσμου. Δεν είναι έτσι και το έχουν αποδείξει. Το έχουν αποδείξει ξεκάθαρα. Οι χρηματαγορέ δουλεύουν για να βελτιώσουν το μερίδιο πλούτου όσων α, λανθασμένα ονομάζονται επενδυτέ. Θα έπρεπε να ονομάζονται κεφαλαιούχοι, καπιταλιστές. Διότι το επενδυτέ έχει θετική χρειά, ενώ το άλλο ε, θα πει ότι απλώ ψάχνουν το κέρδο. Κανένα φιλελεύθερο δεν θα έπρεπε να ψάχνει αυτού του είδου ε, του ε, τους ε, άπλιστους σε σχέση με το κέρδος. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ε, πώς θα γίνει αυτή η ένταξη στο ενωσιακό δίκαιο, διότι απλώς θα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Σα στείλαμε λοιπόν τροπολογίε που υπενήσονται το τι θα έπρεπε να είναι η σωστή νομοθετική ένταξη, αν γινόταν σωστό. Πρώτα απ' όλα, Πρέπει να αλλάξει νομική βάση. Μόνο και μόνο για να βεβαιωθούμε ότι τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου διασφαλίζονται. Νομίζω ότι πολλέ επαναστάσει ξεκίνησαν με το σύνθημα Καμία φορολογία χωρί εκπροσώπηση. Εδώ έχουμε μια δημοσιονομική διαδικασία η οποία όλο και λιγότερο, μα όλο και λιγότερο, ε, έχει να ενταχθεί στο σύστημα δημοκρατικής λογοδοσίας. Τα διορθωτικά μέτρα έπειτα. Εάν έχουμε κάποιο έλλειμμα, κάποιο επικίνδυνο έλλειμμα στον προπολογισμό και αυτά μπορεί να συμβούν, είναι πράγματα που μπορεί να συμβούν και είναι επικίνδυνα για την νομισματική ένωση και για ένα κράτος. Ε, τι διορθωτικές δράσεις, ε, διορθωτικά μέτρα μπορεί να, προ, να, λάβει κανείς. Σε ένα κόσμο όπου τα φορολογικά συστήματα ανταγωνίζονται τα κοινωνικά, προφανώς το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να ισοπεδωθούν οι κοινωνικές δαπάνες και αυτό να πλήξει την ε, αγορά και να καταστραφεί η αγοραστική δύναμη των ενοικιαστών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι λοιπόν να αναλάβει κανείς ε, την δημοσιονομική του ευθύνη μέσα από προγράμματα υποτελεσματικά. Η λιτότητα. Η λιτότητα εντείνει τις, ε, και οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος να εφαρμοστούν ε, προγράμματα κοινωνικής ε, διόρθωσης. Το, έδειξε αυτό η Φινλανδία στις αρχές της ε, δεκαετίας του 90. Μπορεί λοιπόν να προσφέρει ο καθένα το μερίδιο του στην αγορά και οι μετοχοί να κοιτάζανε να συνεισφέρουν στο χάλι που δημιούργησαν με την οικονομική κρίση, λόγω των μετοχών τους. Θα είχαμε πολλά να κερδίσουμε αν έβαινε αυτό, αλλά δεν έχει γίνει όσο για τους ανεξάρτητους φορείς. Διορθωτικά μέτρα. Ε, τα διορθωτικά μέτρα θέλουμε να είναι κοινωνικός και περιβαλλοντικός ε, σχεδιασμένα. Το ίδιο και ανεξάρτητοι φορείς. Είναι ανεξάρτητοι. Βεβαίως μπορεί να έχει κανείς ανεξάρτητους φορείς ε, εάν κάποιος δεν έχει προσχώρηση σε κάποιο κόμμα. Αλλά μπορώ και να κατασκευάσω και ανεξάρτητους φορείς που βασίζονται στο μοντέλο τη νεοκλασικής οικονομία. Δεν ξέρουμε καθόλου πώ μπορεί να λειτουργούν. Μάλιστα, η νεοκλασική θεωρία στην οικονομία είναι παραμύθι, είναι ανέκδοτο. Είναι πραγματικά το κατεξοχήν παράδειγμα ψευδών ειδήσεων, ψευδεπιστήμη. Εδώ λοιπόν θα μπορούσα να ανεχθώ και να δεχθώ ε, ε, έναν δυο ψευδεπιστήμονες, Όμως θα τους πέταγα ε, στην πραγματική οικονομία να κολυμπήσουν στα βαθιά το ίδιο και να συζητήσουν με ανθρώπους που ξέρουν την πραγματική οικονομία και τα προβλήματά της. Ε, αυτή λοιπόν η ε, ανεξάρτητη φορές, τι να πω, καλή τύχη τους εύχομαι. Να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την νομισματική μα ένωση, αλλά αυτά που έχουμε επιτάπητο ούτε κατά διάνοια δεν πλησιάζουν σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Πρόεδρο, ναι, φαίνεται ότι έχουμε πολύ χρόνο αυτή την βραδιά, αλλά πέντε λεπτά και, ε, για τον εισηγητή και τρία για τους υπόλοιπους αν γίνεται. Αν θέλετε να μιλήσετε βέβαια περισσότερο, έχουμε τον ε, χρόνο. Δεν βλέπω εδώ κανέναν. Α, η Μαρίζα Ματίας για τους πρασίνους. Για την ΚΟΕ, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ, θα μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εμείς υποβάλαμε τροπολογία για να απορριφθεί η ένταξη του κανονισμού αυτού στο ενωσιακό δίκαιο. Κυρίως γιατί έχουμε και εμείς συγκεκριμένου πολιτικούς στόχους, συγκεκριμένη πολιτική βούληση. Είναι γνωστή η θέση μας από καιρό. Πιστεύω όμως ότι ακόμη και αυτοί οι συνάδελφοι που ήταν υπέρ της έγκρισης της δημοσιονομικής συνθήκης των εργαλείων που αυτό προβλέπει και των μέσων που προκύπτουν βλέπουν σήμερα με όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια ε, με τις συνέπειες που ζήσαμε ε, τι προκάλεσαν τα μέτρα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας, τις πολιτικές μας αποφάσεις σε ιδεολογικές ε, θεωρίες Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφύγουμε την αιμονή την ιδεολογική, τις τυφλώσεις μας αυτές. Ε, κάποιες φορές κάνουμε το ίδιο σφάλμα ξανά και ξανά. Πρέπει να γίνει μια πραγματική αποτίμηση των ε, επιπτώσεων της δυσμονομικής συνθήκης. Δεν είναι δυνατόν να μην παρατηρήσουμε εδώ ότι τα θεμέλια ε, είναι αμφισβητούμενα. Και εδώ υπάρχει θέμα συντονισμού των κρατών μελών. Ο συντονισμό αυτό να υπάρξει. Αλλά όχι με αυτού του κανόνε που προτείνονται εδώ. Όχι με του κανόνε που έχουμε πει και στο παρελθόν δεν έχουν κανένα επιστημονικό έρισμα. Κανόνε που είναι εντελώ αυθαίρετοι και στην εφαρμογή του. Ε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει. Γιατί για κάποιου η επιβολή είναι πολύ αυστηρή και η εφαρμογή πολύ αυστηρή και για άλλου πολύ επική. Θα πρέπει επίση να δούμε τι γίνεται με του ανεξάρτητου φορεί. Τι γίνεται εδώ. Ε, δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός προσώπου, μιας οντότητας που θα περιοριστεί σε δημοσιονομικές ευθύνες και ε, αρμοδιότητες. Δεν θα ήταν τόσο κακό αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι φορέας ο οποίος θα επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα σε κυβερνήσεις που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μέτρα τα οποία δεν έχουν καν νομιμοποίηση δημοκρατική. Άρα, τι αποτελέσματα θα έχουν. Ε, τα αποτελέσματα πρέπει να τα ζήσει ο κόσμο παρόλα αυτά. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ έρχομαι από μια χώρα που έχει υποφέρει από τι συνέπειε των πολιτικών τη Τρόικα, των πολιτικών προσαρμογή που επιβλήθηκαν και την ιδεολογική επιβολή και αιμονή στην λιτότητα. Εάν όμω θέλουμε να έχουμε κάποια οικονομική ανάπτυξη και να δοθεί κάποιο περιθώριο στην ε, χώρα μου, θα πρέπει να δούμε κριτικά τις προτάσεις που γίνονται εδώ ε, και τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής συνθήκης ε, και το ότι προκάλεσαν. Νομίζω λοιπόν, απλή εντυμότητα, ότι Εάν δούμε τα αποτελέσματα της νομοθεσίας που τώρα έχουμε εφαρμόσει με τη διακυβερνητική συνθήκη, ε, παρατηρούμε ότι όχι απλώς έχουν προκληθεί μακροοικονομικές ανισορροπίες και ανισότητες, αλλά και κοινωνική κρίση. εδώ λοιπόν Κάπω θα πρέπει να σταματήσουμε, να πάρουμε βαθιές ανάσες, να σκεφτούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λογική λύση. Γιατί πάει έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως για τα πολιτικά μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες είτε της οικονομίας της Ευρώπης είτε στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων που περιμένουν κάτι από την Ευρώπη. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν α σταθούμε δύο λεπτά, να πάρουμε δύο ανάσει, να σκεφτούμε ποια είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα που χρειαζόμαστε, διότι δεν είναι αυτή που μα προτείνεται. Εάν δεν ε, σκεφτούμε τι θα κάνουμε από την αρχή, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε προ τα μπρο ε, ε χωρί να κοιτάζουμε ε, που πάμε. Πρέπει να δώσουμε ένα σωστό μήνυμα συντονισμού στον πολιτικό τη δημοσιονομική πολιτική τη Ευρώπη, κάτι που δεν έχει γίνει ω τώρα. Αυτό που ω τώρα έχει γίνει είναι η ιδεολογική ε, αιμονή, η τύφλωση αυτή και η ε, πεισματική εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στο Catch the Eye. Κυρία Μπερές. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή έχει ενδιαφέρον. λόγω του ότι η οικονομική πολιτική εξελίσσεται με τον τρόπο που γνωρίζουμε, δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες να εκφραστούμε από αυτές. Τρεις παρατηρήσεις λοιπόν. Η πρώτη ακούστηκε ήδη, αλλά μπορεί ο καθένας νομίζω να το πει έτσι ώστε το μήνυμα να ακουστεί καλά. Κανένας πια σχεδόν στην Ευρώπη δεν θεωρεί ότι το σύμφωνο σταθερότητας αποτελεί το σωστό πλαίσιο στο εσωτερικό της ζώνης ευρώ. Ίσως κάποιοι να το πιστεύουν, αλλά είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί όταν βλέπουμε ότι αυτό οδηγεί συστηματικά σε εκλογή του Σαλβίνη, ας πούμε, ε, κάτι σημαίνει ε, αυτό ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορούμε λοιπόν επίσης να δίνουμε δήθεν την εντύπωση ότι προχωράμε σε νομικό επίπεδο χωρίς να θέτουμε το ε, ζήτημα το οποίο τίθεται που είναι η ένταξη της ε, δημοσιονομικής συνθήκης την οποία πάντα απορρίψαμε σε, κοινωνικό, σε κοινοτικό επίπεδο και το είπε και ο Φίλιπ Λάμπερτ πάντα πιστεύουμε εμείς ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε με μια σοβαρή αξιολόγηση η αξιολόγηση αυτή σοβαρή γίνεται τώρα και υπάρχει θέμα δημοσιονομικό το οποίο συνδέεται με την συζήτηση για το Σύμφωνο Σταθερότητας, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα η συζήτηση αυτή. Υπάρχει επίσης και άλλο ένα θέμα το οποίο ακούω συχνά και το οποίο τι λέει, ότι σε επίπεδο θεσμικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί διαβουλευτικά και μόνο, οπότε απλά θα πρέπει να είναι ευγενέ και να μπορεί να συμμετέχει ελαφρά στη συζήτηση. Δεν έχει νόημα αυτό. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τέτοιου είδου επιχειρήματα και από τη δική μου πολιτική ομάδα και από τη δική σα κυρία Χούμπνερ, όταν νομοθετούσαμε για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Ότι θα έπρεπε να ήμασταν soft, ότι δεν θα έπρεπε να απορρίπταμε εμείς για έναν και μόνο λόγο νομικό ή ε, οικονομικό. Κοιτάξτε, όλα τα έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την πραγματικότητα των διαπραγματεύσεων και γι' αυτό είναι σημαντικό να μην τροποποιήσουμε τη νομική βάση γιατί αυτό θα καταστήσει πολύ εύθραστες τις συζητήσεις λόγω των στόχων των πολιτικών τους οποίους έχουμε μπροστά μας και θα πρέπει να καταστήσουμε τους στόχους αυτούς συμβατούς με τομείς όπως η αηφόρος ανάπτυξη, κάτι το οποίο δυστυχώς μέχρι τώρα στην πλαίσιο αυτό συζήτησης δεν γίνεται. Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημοσιονομική συνθήκη πρέπει να το θυμίσω, ήταν απόκριση, μια απόκριση έκτακτη στην κρίση των ε, κρατικών χρεών και ελλημάτων. Ήταν μια διακυβερνητική λύση στο περιθώριο των όσων μέχρι τώρα προβλέπονταν στην Ένωση και τα συμβαλόμενα μέρη, τα κράτη δηλαδή, είχαν συμφωνήσει τότε ότι θα υπάρξει μελλοντική ένταξη των κανόνων της δημοσιονομικής συνθήκης στο ενωσιακό δίκαιο. Και ότι αυτό βέβαια θα έπρεπε να ε, ακολουθήσει μια αξιολόγηση της εμπειρίας και της αποτίμησης της εφαρμογής της συνθήκης. Άρα και ενδεχόμενη αναθεώρηση των κανόνων αυτών. Το να λέμε τώρα ότι αυτοί που απορρίπτουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ζητά απλώ ένταξη τη δημοσιονομική συνθήκη ε, στου ευρωπαϊκού κανόνε, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα πει ότι το κοινοβούλιο αυτό στηρίζει διακυβερνητικέ ε, συνεννοήσεις και εξέβρεση λύσεων, είναι πολιτικό ψεύδο. Αυτό που απορρίπτει το κοινοβούλιο αυτό στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επειδή, ότι απαιτεί μάλλον, ο λόγο είναι ότι απαιτεί να αξιολογήσουμε το τι ζήσαμε μετά την εφαρμογή τη δημοσιονομική συνθήκη και όπου χρειάζεται να αναθεωρηθούν κανόνες. Κάτι που προβλεπόταν και στην προηγούμενη, την ίδια την δημοσιονομική συνθήκη, στην αρχική της μορφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει διακυβερνητικές λύσεις να καθαγιαστούν και να καθιερωθούν, αλλά να ε, κοιτάξουμε μετά την εμπειρία που ζήσαμε με την κρίση των κρατικών χρεών, μετά την, ε, τα βιώματα της πολιτικής κρίσης των τελευταίων ετών, τη σύγχυση που σήμερα υπάρχει σε σχέση με την ερμηνεία των κανόνων. Κάθε φορά που υποβάλλει κανείς ένα σχέδιο προπολογισμού, κράτη, κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και το Συμβούλιο, τα ανεξάρτητα Συμβούλια Δημοσιονομικής Πολιτικής, δεν μπορούν πια να συνεννοηθούν. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η εφαρμογή των κανόνων στην πράξη. Άρα τι σημαίνει αυτό. Έχουμε άπειρους λόγους να κάνουμε μια αναθεώρηση. Και μάλιστα με, όσο πιο σύντομα γίνεται, με σοβαρότητα, να δούμε τι διορθώσεις και αναθεωρήσεις χρειάζονται, ώστε να έχουμε και ένα δίκαιο της Ένωσης που να μπορεί να δώσει δημοσιονομικές πολιτικές αποκρίσεις, πραγματικό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και όλα αυτά να βρισκόνται στο ύψος των προσδοκιών των πολιτών. Thank you. I Ευχαριστώ. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Η κυρία Χιούμπνερ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ε, έγινε αυτή η συζήτηση για όλο το δημοσιονομικό πλαίσιο, τα νομοθετικά, τις δέσμες νομοθετικών μέτρων κλπ. Ε, νομίζω όμως ότι συζητάμε πράγματα που ε, ανήκουν σε διαφορετικά θέματα. Εδώ έχουμε την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους του άρθρου 3. Αυτό δεν δημιουργεί νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτε αλλάζει ε, τις τα ε, δέσμες νομοθετικών μέτρων που λέγονται εξάπτυχο και δίπτυχο. Ο, ο στόχος είναι διαφορετικός και μπορεί να συσχετιστεί προς τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου από παλιά σχετικά με την ε, μεταφορά αυτής της συνθήκης στην ένωμη τάξη της Ένωσης. Γιατί ε, κάποιος ανεξάρτητος ε, κάποιο, κάποιο ανεξάρτητο μέσον ε, για να ενσωματωθεί μπορεί, ε, αν είναι ανεξάρτητο, ε, μπορεί να αλλάξει τελείως το περιεχόμενό του και αυτό να επηρεάσει την πολιτική της Ένωσης στο δημοσιονομικό επίπεδο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την οδηγία για να αλλάξετε άρδιν το πλαίσιο, αυτό σε νομικό επίπεδο δεν γίνεται. Γι' αυτό και η τροπολογία σας δεν προτείνει αυτή την αλλαγή. Ε, ε, θέλετε να στείλετε ένα πολιτικό μήνυμα για να εκφράσετε το θυμό σας και την ε, βούλησή σας να εργαστείτε ουσιαστικά πάνω στο θέμα. Εδώ όμως έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Αν δεχτούμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση, τότε η οδηγία δεν θα συνάδει με το υπόλοιπο πλαίσιο που δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε έτσι κι αλλιώς μέσα από αυτή την οδηγία. Γι' αυτό αυτή η οδηγία εν μέρη μόνο, τροποποιεί, ε, ε, εν μέρη ενσωματώνει κάτι που δεν είχε ε, ενσωματωθεί, ή ολοκληρωθεί, αλλά δεν κλείνει καμιά, ντόρα, καμιά πόρτα, συγγνώμη, ούτε άπτεται αυτών των θεμάτων που θε, βάζετε εσείς τώρα. Γι' αυτό μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα έχουμε και την αναθεώρηση, την επανεξέταση του χρόνου των ε, νομοθετικών μέτρων 6 και 2. Αυτό είναι διαφορετικό όμως. Γι' αυτό προτείνω να κάνουμε αυτά που υπάγονται σε αυτή την οδηγία και σε αυτή την μεταφορά στην ενωμητάξη της Ένωσης. Δεν μιλάμε εδώ για αλλαγή της συνθήκης. Μιλάμε για αυτό που βρίσκεται στο πλαίσιο που δεν έχει ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Προτείνω να κάνουμε μια συζήτηση με τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, παρόλο που εδώ δεν επιδέχονται τα θέματα αυτά πολλών συμβιβαστικών λύσεων. Μπορούμε να κάνουμε μια συνάντηση με όσους ενδιαφέρονται να το συζητήσουμε αυτό περισσότερο αλλά επειδή ε, ζούμε από ό,τι φαίνεται σε διαφορετικούς κόσμους σε ό,τι αφορά το, το, το νόμο, την νομοθεσία, ε, ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Πάντως εγώ είμαι πρόθυμη να το συζητήσω. Το, πάνω το δω θετικά. Συμφωνώ μαζί σου σε πολλά όπως γνωρίζεις πολύ καλά, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα δεν πρέπει να ε, μπερδέψουμε τους δύο στόχους. Είναι διαφορετικός ο στόχος που αφορά αυτό το μικρό κομμάτι της συνθήκης και άλλο αυτό που λες εσύ που θέλεις μια θεμελιώδη ε, παρεξέταση. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτε από αυτά που θέτεις εσύ εδώ εν προκειμένου. Δεν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Όσοι ασχολείστε με το θέμα, πάτε στη συνάντησή της Τετάρτης να δείτε τι μπορεί να γίνει. Ε, στις 27 Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ για το θέμα αυτό. Ε, ευχαριστώ για την προσοχή σας και προχωρούμε στο τελευταίο θέμα μας. Η ε, τήσια ε, έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κυρία Κάπελ, η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι σχεδόν 9.30. Κάναμε πολύ εντατική συζήτηση και ξαναγυρίσαμε στο πρόγραμμά μας όπως το είχαμε ενδεικτικά. Ε, ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Υπάρχουν πολλές, πολλές τροπολογίες. 165, 30% παραπάνω από πέρσι. Γιατί, διότι επειδή είναι μικρή η έκθεση, δεν είχαμε πολύ δυνατότητα να ε, επεκταθούμε στο κείμενο. Γι' αυτό ευχαριστώ, στου, ευχαριστώ τους σκιώδες για τις ε, παρεμβάσεις τους που βοήθησαν να κάνουμε την έκθεση εκτενέστερη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Και εγώ κατέθεσα μια σειρά τροπολογιών. Με, τη, με το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών Προσθέσαμε τρία νέα κεφάλαια, τα οποία καλύφθηκαν από τις τροπολογίες. Είναι η φορολογική συμμόρφωση, η εντολή εξωτερικού δανεισμού και η διαφάνεια. Συνολικά έχουμε εννέα συμβιβαστικές, τρεις τις ανέφερα, που καλύπτουν 15 άρθρα της αρχικής έκθεσης. Πολλά άρθρα δεν είχαν δε, ε, τροπολογίες. Ε, υπήρχε συμφωνία στους περισσότερους τομείς, σε τεχνικό επίπεδο μπορέσαμε να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε καλά και το πρωί είχαμε τελευταία τεχνικής φύσεως συνάντηση, έχουμε ε, ε αύριο 8 το πρωί ε, συνάντηση για να συμφωνήσουμε και την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί στην έκονη έκθεση. Αύριο ελπίζω να συμφωνήσουμε, είμαι αισιόδοξη και περιμένω με χαρά την αυριανή συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Κάπελ. Δεν έχω κανέναν εδώ από το ΕΛΚ. Την ομάδα μου, ο Σάντερ Λούνες, δεν μπόρεσε να έρθει. Δεν θα ήθελα να αναφέρω ότι χάρη στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, τις προσπάθειες ε, του κυρίου Λούνες στα τελευταία χρόνια, ε, ε, τώρα είναι υπουργό Άμυνα στο Βέλγιο. οπότε ως συντονίστρια δεν μπόρεσα να τον αντικαταστήσω, δεν πρόλαβα. Δυστυχώς δεν βλέπω κάποιον λοιπόν και δεν βρήκα κανένα. Ο κύριος Παπαδημούλης όμως ε, ζήτησε το λόγο από την ομάδα Γκουε. Ε, σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω εκ μέρους και όχι μόνο της πολιτικής μου ομάδας, αλλά ενδεχομένως και άλλων σκιωδών εισηγητών που δεν είναι σήμερα παρόντες. Ε, νομίζω ότι ένας από τους λόγους που έχουμε καταθέσει σε αυτή την έκθεση που μας παρουσίασε η συγγήτρια πολύ περισσότερες τροπολογίες από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές δεν είναι μόνο το μικρό μέγεθος της έκθεσης αλλά και μία μειωμένη διάθεση μέχρι τώρα από την εισηγήτρια να ενσωματώσει παρατηρήσεις και προτάσεις που έχουμε καταθέσει εδώ στη διάρκεια της συζήτησης γιατί υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ανάγκες που δεν μπορούμε να τις κρύβουμε κάτω από το χαλί, γράφοντας απλώς μία έκθεση για την ιστορία του πώς ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και είμαστε σε μια φάση που χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξους στόχους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποτελεσματικότερη στοχοθεσία των επενδύσεων να πάνε περισσότερο οι επενδύσεις στις περιφέρειες που τις έχουν περισσότερη ανάγκη, που είχαν την μεγαλύτερη επένδυση στα χρόνια της κρίσης, που είχαν την υψηλότερη ενεργεία, μεγαλύτερη διαφάνεια στις αποφάσεις, ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, ενίσχυση των πολιτικών συνοχής και μέσα από τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε συνδυασμό με τις πολιτικές συνοχής και να πάρουμε περισσότερο υπόψη μας και τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θέτει εν ώψη του 2030 ο ΟΗΕ. Θέλουμε δηλαδή μέσα από την έκθεση να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων περισσότερες φιλοεπενδυτικές πολιτικές για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρότερη μέρημνα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το περιβάλλον, την καινοτομία. Και εδώ υπάρχει ανάγκη να φύγουμε από τη λογική του business as usual. Ιδιαίτερα για περιοχές που υποφέρουν από μακροχρόνια ανεργία, νεανική μετανάστευση και ελλείμματα κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής. Αύριο το πρωί στις 8 η ώρα ε, θα έχουμε ένα ακόμη shadow meeting, εμείς θα προσέλθουμε με θέσεις και προτάσεις, γιατί πιστεύω ότι οι μέχρι τώρα προσπάθειες της εισηγήτριας για συμβιβαστικές προτάσεις δεν είναι επαρκής και ευελπιστώ ότι οι προτάσεις μας οι παρόμοιες προτάσεις θα υποστηριχθούν και από ε, υπόλοιπους και από άλλους κοιόδης εισηγητές άλλων πολιτικών ομάδων που σήμερα δεν είχαν την ευκαιρία να είναι παρόντες. Ευχαριστώ. With that, I'd like to hand back to the rapporteur for closing remarks. Mrs. Cabell. Η συγκεκριά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Παπαδημούλη για την τοποθέτησή του και ελπίζω ότι αύριο θα είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα για όλους ούτως ώστε την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση. Thank you. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αύριο η Σκιώδης και 19-20 Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία. Αυτή είναι, αυτό ε, ε, ε, είναι το πρόγραμμα. Ε, το σημείο 10 είναι τα διάφορα. Δύο μέλη βρίσκονται παρόντα αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχουν να πούν τίποτα, κλείνουμε τη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι 19 Νοεμβρίου 3 με 6.30. Είναι Δευτέρα. Και Τρίτη 20 Νοεμβρίου μεταξύ 9 και 12.30 και από 2.30 μέχρι 6.30. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.